course. Uh, uh, uh, ορίσατε στη συνεδρίαση αυτή μεταξύ Επιτροπών Απασχόλησης ε, και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Παιδείας. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσης διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, Συμφωνείτε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, ναι. Διερμηνία σήμερα έχουμε και από τα ελληνικά μεταξύ άλλων. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Θα ξεκινήσουμε με τις συζητήσεις ε, για τις καλύτερες υπηρεσίες, ε, για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα. Να πω λοιπόν ε, δύο λόγια για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς ε, χαίρομαι που καταφέραμε να κανονίσουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση μεταξύ των δύο επιτροπών ε, της Επιτροπής Πολιτισμού και της Επιτροπής Απασχόλησης και θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Πολιτισμού εδώ σήμερα. Πολλά κοινά ενδιαφέροντα έχουμε. Ε, όσον αφορά το όσα συζητώνται στι επιτροπέ μα αυτή τη στιγμή, αλλά και ανέκαθεν. Ανέκαθεν συζητούσαμε, θα έλεγα, τι δεξιότητε. Σήμερα θα συζητήσουμε μια πρόταση τη Κομισιόν για ένα εξυγχρονισμένο πας και θα ανταλλάξουμε απόψεις για το θεματολόγιο δεξιοτήτων ε, στην Ευρώπη. Να σας υπενθυμίσω ότι τα δύο αυτά αρχεία θα ε, μας απασχολήσουν δυναμή του κανόνα το άρθρο 55, αυτό σημαίνει ότι ο καθένα ε, εισηγητή ε, από την κάθε επιτροπή θα συντάξει μία έκθεση που θα ψηφιστεί. Θα συναντιόμαστε λοιπόν μέχρι τον Ιούνιο τακτικά. Υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε από κοινού, που μας ενδιαφέρουν από κοινού, οπότε θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε και κοινέ θέσεις για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεδομένων αυτών, να δώσω το λόγο στη νέα πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού, την κυρία Κάμερβερτ. Έχετε το λόγο. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να σας χαιρετήσω από τη δική μου πλευρά και θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Απασχόλησης η οποία μας υποδέχεται εδώ και κάνουμε την κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Πολιτισμού και μπορούμε να έχουμε αυτή την κοινή συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς εμπλέκει και ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τις δύο Επιτροπές. Μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα να προωθήσουμε αυτό το θέμα στην, ε, στο θεματολόγιο αυτό λοιπόν της ικανότητας και έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι το πλαίσιο αυτό το οποίο υπάρχει για τις δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί ήδη μια αναθεώρηση. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας μας έχει οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πρέπει λοιπόν να ευγεροποιηθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των χρηστών και επίσης να έχουμε και μια καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση, ακόμα και την άτυπη, τις άτιμες μορφές ε, εκπαίδευση και κατάρτιση και όλα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε συνάφεια με τις δυνατότητες απασχόλησης και επομένως εναπόκειται σε εμά να αξιολογήσουμε υπό αυτό το πρίσμα την πρόταση της Κομισιόν. Φυσικά υπάρχουν και κριτικές απόψεις για μας για το Europass. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο είχε σαν στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν δεξιότητες και προσόντα. Ο στόχος μας όμως θα πρέπει να είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με πιο καινοτόμο τρόπο και επομένως να λάβουμε υπόψη μας τις τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες ε, λαμβάνουν χώρα και να μπορέσουμε να παραμείνουμε στο ύψος των καιρών να μπορέσουμε να κάνουμε τι απαραίτητε λοιπόν τροποποίησει στο σύστημα Europass. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ξαναδίνω το λόγο στην πρόεδρο τη Επιτροπής Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα όσα είπατε εν είδη αγωγής. Πράγματι υπάρχει ανάγκη να εξυγχρονίσουμε τα εργαλεία και τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με την Επίτροπο Τάισεν είχαν μία συζήτηση σχετικά στην ε, Ολομέλεια στο Στρασβούργο και δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε. Ε, συμμετείχαν μέλη και των δύο επιτροπών, αλλά και, άλλα, και άλλοι συνάδελφοι από άλλες επιτροπές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι ε, θα ε, φαίνονται οι ανάγκες που υπάρχουν της αγοράς εργασίας ε, σε όλους τους ενδεχόμενους χρήστες, ειδικότερα όσον αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης και ότι πρέπει να, πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή σύμφωνα με τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Πρέπει να μπορούν τα εργαλεία να υποστηρίζουν και τους εργαζόμενους, αλλά και τους μαθητευόμενους κατά τη διάρκεια της επαγγελματική του ζωής. Πολλές φορές χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα πράγματα παραπάνω από μία φορά στη ζωή μας και δεν χρειάζεται να το κάνει κανείς όταν ξεκινά την ενήλικη ζωή του ε, αλλά πολλές φορές μέσα ε, στην ε, μετέπειτα ζωή του. Φαντάζομαι ότι οι συνεισηγητές θα καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό που θα είναι αποδεκτός από όλους και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαλίνοφ, που είναι ο εισηγητής εξ ονόματος Επιτροπής Πολιτισμού και μετά στον κύριο ΜΑΜ, που είναι ο εισηγητής της Επιτροπής Απασχόλησης. Πέντε λεπτά έκαστος. Κύριε Μαλίνοφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, θα σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο ε, σε μένα πρώτο. Ο κύριος ε, Μαν θα παραθέσει και εκείνος πολύ σημαντικά επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση γιατί υπήρξε μια συνεννόηση μεταξύ μας. Θα επαναλάβω όπως είπατε και εσείς ότι υπάρχει μία επίγουσα ε, ανάγκη ε, ανανέωσης, γιατί ό,τι και να πούμε για το Europass, ε, ό,τι στοιχεία και αν δώσουμε, πόσο επιτυχημένο είναι, πόσο γνωστό είναι, πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί, τα έγγραφα Europass έχουν, έχουν παραμείνει ίδια εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ο κοινό παρονομαστή που αποδέχονται όλοι ε, και τα κράτη-μέλη και διάφοροι εμπλεκόμενοι φορεί ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ανανέωση. Όμω ε, για να ε, είναι όσο το δυνατόν χρησιμότερη αυτή η ανανέωση θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι έχουν εκφραστεί πολλέ ανησυχίε από πολλά κράτη-μέλη, περισσότερα από αυτά που χρειάζονται για οποιαδήποτε διαδικασία κίτρινη κάρτα ή οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. Αυτέ οι ανησυχίε εμφανίστηκαν εγκρίθηκαν σχεδόν αμέσως και ε, δείχνει ότι υπάρχει μία συνένεση επί κάποιων σημείων και επειδή δεν θεωρεί κανείς ότι υπάρχει καμία συνωμοσία εναντίον της ε, αναθεώρησης ε, του Europass πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτές τις ε, ανησυχίες γιατί τα επιχειρήματα είναι πολύ σωστά και ακόμη και εγώ που ήμουν έτσι πιο ρίσοσπαστικός ως προς την προσέγγιση μου μπορώ να καταλάβω τα επιχειρήματα αυτά. Η πρόταση δεν ήταν πάρα πολύ σαφής και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλά ερωτήματα σε πολλά προβλήματα σε πολλές χώρες. Ε, αυτές ε, οι ανησυχίες λοιπόν είναι πολύ σημαντικές και με απασχολούν και εμένα. Είμαι σίγουρος ότι και ο κύριος Μαν θα προσθέσει και άλλα επιχειρήματα. Όσον αφορά τον ε, τίτλο εργασίας, αναθεώρηση του Europass, αν διαβάσει κανείς ε, την πρόταση είναι πολύ πιο έλευθη. Ε, αναφέρονται μεταξύ των προθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρόκειται για ένα νέο μέσο. Οπότε η πρώτη ανησυχία είναι ότι το Ευρώπας πρέπει να εξυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στι ανάγκε των χρηστών, αλλά δεν πρέπει να ε, αποτελέσει ένα εντελώ νέο μέσο. Η διατύπωση της ε, παλαιάς νομική βάσης πρέπει να χρησιμεύσει ως καθοδήγηση. Ε, Λαμβανωμένη υπόψη της μεγάλης κλίμακας αυτής της πρότασης για ένα νέο Europass, οι τεχνικές πτυχές χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων όπως και περισσότερων πληροφοριών για το κόστος ανάπτυξης του συστήματος. Υπάρχει γενική συνένεση ε, σε σχέση με ε, την ταξινόμηση ε, ΕΣΚΟ, την ταξινόμηση ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς, δεν έχει ολοκληρωθεί. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρότασης είναι πρόημο. Υπάρχει γενική συνένεση ότι θα έπρεπε να διαγραφεί εντελώς από την πρόταση. Μία ακόμη ανησυχία αφορά τις ομάδε εμπειρογνωμόνων που θα υποκαθαστήσουν ε, τους εμπειρογνώμονε ε, που ασχολούνται με τα θέματα προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωση. Πρέπει να είναι σαφέ ότι το Europass ε, δεν θα έχει σκοπό να αλλάξει το σύστημα που υπάρχει στα κράτη-μέλη, παρά το γεγονός ότι αυτός ο φόβος έχει εκφραστεί πολλές φορές στα διάφορα έγγραφα που έχουν ε, εκφράσει την άποψη των κρατών μελών. Προσπαθώ να συνοψίσω τις βασικές ανησυχίες, δεν θα ε, αναφερθώ στις δικές μου, προσπαθώ να αναφερθώ γενικά σε αυτούς τους φόβους και τις ανησυχίες που εξηγούν τις επικρίσεις ε, επί, τις ε, των οποίων συμφωνούν ε, τα κράτη-μέλη που εξέφρασαν αντιρρήσεις. Όσον αφορά τώρα την ολοκλήρωση εντολή όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων ε, για την αναθεώρηση των, ε, ε, του Europass και την αντικατάσταση αυτών σε επίπεδο Ένωση. η πρόταση αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνει υπόψη τις διάφορες εθνικές δομές και τις ανάγκες των κρατών μελών και δεν δίνει καμία ευελιξία από ό,τι φαίνεται όσον αφορά την εφαρμογή του νέου συστήματο. Μία ακόμη ανησυχία αφορά το ρόλο των κρατών μελών και ε, το αίτημα δημιουργίας νέων ε, ε, κέντρων συντονισμού στα κράτη-μέλη εθνικών. Αυτό είναι δύσκολο γιατί το να υπάρξει χρηματοδότηση για αυτό έρχεται σε αντίθεση, παρεμβαίνει στις εθνικές αρμοδιότητες και στις ε, αρμοδιότητες των κρατών μελών ε, σε σχέση με την οργάνωση των δικών του συστημάτων. Θα σταματήσω εδώ. Σε γενικές γραμμές συμφωνούν όλοι ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης, ε, ότι το Europass όντως ήταν επιτυχές, ότι χρειάζονται τώρα κάποιες αλλαγές, όμως... Είναι πολύ φιλόδοξο ε, απαιτεί πολλές αλλαγές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η ε, γενική μου προσέγγιση. Ίσως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη, ειδικότερα όλα αυτά τα σημεία ε, για τα οποία τα 14 κράτη-μέλη έθεσαν, εξέφρασαν κάποιες αντιρρήσεις που αφορά για παράδειγμα το γεγονός ότι το ΕΣΚΟ, αυτή η ταξινόμηση των προσόντων ε, πρέπει να αποκλειστεί από την πρόταση. Αλλά ελπίζω ότι θα υπάρξει ένας συμβιβασμός για την τελική εκδοχή του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Είναι δύσκολα να μην συμφωνήσει κανείς ε, καθαρά Δευτέρα για αυτά τα θέματα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος αν υπάρχουν διαφορές απόψεων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δούμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε καλύτερα για να δούμε πώς πρέπει να κατευθύνουμε τα θέματα αυτά του Europass. Το Europass βέβαια είναι κάτι το οποίο έχει ακολουθήσει μια σωστή κατεύθυνση, θέλει να πετύχει ένα σωστό ρόλο. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτή την ιδέα. Το θεματολόγιο αυτό υποστηρίζεται πλήρως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βασικά θέλουμε να εξυγχρονίσουμε το εργαλείο αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το εργαλείο, απλώ θα πρέπει να το ενημερώσουμε και να το επικαιροποιήσουμε ώστε να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στι νέε προκλήσει. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω απόλυτα αυτά τα οποία λέει ο κύριο Μαρινόφ. Ενώ κάποια κράτη-μέλη έχουν διατυπώσει αντιρρήσει και αμφιβολίες για τα θέματα αυτά. Είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι στα κράτη-μέλη υπάρχουν ορισμένα εργαλεία τα οποία λειτουργούν, γι' αυτό υπάρχει και μια δυσπιστία σε σχέση με ένα νέο εργαλείο. Φοβούνται να μην υπάρξουν περαιτέρω γραφειοκρατικά εμπόδια. Είναι απαραίτητο λοιπόν εμεί να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε τα απαραίτητα δεδομένα, <clears throat> να έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασία αυτών των στοιχείων, χωρί όμω περιττό άχθος. Η πρόταση της Κομισιόν λέει ότι ό,τι νέα εργαλεία ε, υπάρχουν θα πρέπει να έχουν ένα εθελοντικό χαρακτήρα. Αλλά είναι κάτι τέτοιο αυτό το οποίο μπορούμε να το δεχτούμε. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να διατηρούν αρμοδιότητα για τον τομέα αυτό και αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί. Ο στόχος λοιπόν του Europass είναι να μπορέσει να υπάρξει μεταφορά πληροφοριών προς το όφελος του τελικού χρήστη αλλά ο στόχος είναι να υπάρξει και σωστή αντιμετώπιση του άχθους και του κόστους αυτού του συστήματος. Αυτό θα μας υποχρέωσει σε ορισμένα σημεία να το κάνουμε πιο υποχρεωτικό το σύστημα Europass. Και εδώ έρχομαι στο θέμα του ΕΣΚΟ για τις ικανότητες και, τις, ε, και τα προσόντα που χρειάζονται. Να μπορεί κανείς να έχει ένα καλύτερο προσανατολισμό των προσόντων αυτών προς, την, προς τις ανάγκες της αγοράς αυτή τη στιγμή. Το ΕΣΚΟ είναι μια πολύ καλή δυνατότητα. Όταν λειτουργεί στο διαδίκτυο δεν οδηγεί σε πρόσθετο κόστος και μπορεί να είναι προσβάσιμο από όλους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η αυτόματη μεταφορά και ε, μετάφραση των ικανοτήτων και των προσόντων από τη μία γλώσσα στην άλλη, ώστε να μπορούν να είναι σαφή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι είναι... Είμαι σύμφωνος με τον εισηγητή σε γραμμές, αλλά θέλω να τονίσω το ότι είναι απαραίτητο να παραμείνει αυτό το σύστημα εθελοντικό, ώστε να μπορεί κάθε χώρα να θέτει τα δικά της κριτήρια σε σχέση με τα προσόντα και να μην προκύψει μια ισοπαίδωση προς τα κάτω. Και υπάρχει και το θέμα της ευκυβερνησίας αυτού του συστήματος. Έχουμε ομάδες με εθνικούς εμπειρογνώμονες που μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλά μεταξύ τους. Κάποιοι από αυτούς φοβούνται όμως ότι θα προκύψει μια έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης ή ικανότητας. Αυτές οι ομάδες εμπειρογνώμων που έχουμε τώρα έχουν αποδείξει την ικανότητά τους, έχουν λειτουργήσει πολύ καλά μέχρι τώρα εμείς ξέρουμε ήδη από την εσωτερική κατάσταση στη Γερμανία ότι είναι απαραίτητο οι διάφοροι φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να συνεργάζονται περισσότερο. Με τον τρόπο αυτό, μονάχα με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει το Europass να γίνει ένα πραγματικό ε, εργαλείο για όλους. Επομένως, είναι απαραίτητο να τονίσουμε τον καλύτερο διάλογο που πρέπει να διαμειφθεί μεταξύ των εθνικών αρχών. Να υπάρξει λοιπόν μια καλύτερη συνεργασία. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά μας στοιχεία πρέπει και πάλι να εξασφαλίσουμε ποια είναι η σωστή κατεύθυνση, σε ποιο βαθμό πρέπει να υπάρχει το εθελοντικό στοιχείο και πού θα πρέπει να υπάρχει και μια υποχρεωτική πτυχή. Και γι' αυτό είναι το έργο και των δύο επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασχοληθούν με το θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση για τα θέματα αυτά. Η συνένεση βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία ήδη λειτουργούν και λειτουργούν πολύ σωστά στα κράτη-μέλη μας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Mann. I'll you. Ευχαριστούμε κύριε Μαν. Θα πω και εγώ δύο λόγια. Αφού είμαι σκιώδης ε, από την Επιτροπή Απασχόλησης ε, εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών για την εκθεσή αυτή. σε γενικές γραμμές ε, ε, χαίρομαι που γίνεται αναθεώρηση του Europass γιατί κάποια ζητήματα κλειδιά που έχουν εμφανιστεί χρειάζονται αναλυτικότερη εξέταση και διόρθωση. Ο κύριος σκοπός ε, του να γίνει το πας πιο φιλικό προς το χρήστη είναι θεμητός, αλλά χρειάζεται και διαφάνεια ώστε να γίνει το πας πιο ελκυστικό για ένα ευρύτερο κοινό. Όπως πολύ ξέρετε, το 60% των ορτιθέντων στην έρευνα που δεν το είχαν χρησιμοποιήσει δεν ήξεραν καν την ύπαρξή του. Το ίδιο ισχύει και για ιδιωτικές εταιρείε, πιθανού εργοδότες που είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τις ε, υπηρεσίες αυτές ε, σήμερα. Οπότε κατά την αναθεώρηση θα πρέπει να μην ξεχάσουμε να αναθεωρήσουμε και αυτό το ζήτημα, να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα. Τώρα η διαφάνεια των δεξιοτήτων που είναι ένας από τους σκοπούς του Europass θα πρέπει να ευξηθεί ε, καθώς ο κόσμος θα γνωρίζει περισσότερο τα εργαλεία και τις υπηρεσίες, ε, όχι μόνο όσοι χρησιμοποιούν ήδη τις υπηρεσίες αυτές. Κάτι άλλο τώρα. Πολλά κράτη-μέλη, όπως αναφέρατε κι εσείς ήδη, καθώς και, καθώς και πολλοί ενδιαφερόμενοι, έχουν εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά τις αλλαγές στο Europass και τη συμπερίληψη νέων εργαλείων. Οι αλλαγές αυτές δεν έχουν παρουσιαστεί καθαρά, οπότε θα απέχω από το να σχολιάσω προς το παρόν. Αλλά θα ήθελα να πω ότι η Κομισιόν θα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα ζητήματα αυτά. Επίσης και εγώ και μέρα με απασχολούν κάποια θέματα όπως ε, η σχέση μεταξύ του Europass ε, και του EQF και του ESCO. Το EQF είναι εθελοντικό και το ESCO εξακολουθεί να βρίσκεται σε πιλωτική φάση. Επίσης παροτρύνω την Κομισιόν να μην αποσύρει τι ομάδε εμπειρογνωμών που σχετίζονται με το Europass, ότι από τη δική μου εμπειρία η συμμετοχή του, η συμβολή αυτών των ομάδων εμπειρογνωμόνων ε, είναι πολύ σημαντική για την υψηλή ποιότητα των εργαλείων και την ευχρηστία των εργαλείων. Αυτά ήθελα εγώ να πω ω παρατηρήσεις ω και Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Σμόλκοβα που εκπροσωπεί τους σοσιαλιστές ε, και την Επιτροπή Πολιτισμού. Α, συγγνώμη, δεν σας είδα. Έχετε το λόγο, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχει διατυπώσει την πρότασή της σε σχέση με τα προσόντα και τις δεξιότητες. Εγώ θα ήθελα να γνωρίσω καλύτερα πώς λειτουργεί το σύστημα Europass και να έχω και προσωπική επαφή με τους εργαζόμενους σε αυτό το κέντρο για το Europass, ώστε να μπορώ να καταλάβω καλύτερα τα θετικά και τα αρνητικά αυτού του συστήματος και πώς μπορούν να βελτιωθούν. Υπάρχει, όπως ξέρουμε, το σύστημα αυτό στο διαδίκτυο, το οποίο μεταφέρει τις ε, προτάσεις για τους ε, εργαζόμενους και τους ε, φυτώντες λοιπά Είναι προς το συμφέρον όλων μας να μπορεί να βελτιωθεί αυτό το σύστημα ώστε να μπορέσει να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες και να προσαρμοστεί σε, μια, ε, σε ένα χώρο εργασίας ο οποίος είναι σε συνεχή ρευστότητα και αλλαγή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει <clears throat> να υπάρξει και διεύρυνση του συστήματος αυτού του Europass και να διευρυνθεί, να διασυνδεθεί με άλλα ευρωπαϊκά συστήματα, όπως αυτό που έχει να κάνει με την αναγνώριση των πτυχίων κτλ. Υπάρχουν βέβαια και οι ανησυχίες που πιστεύω ότι είναι και δικαιολογημένε ότι θα έρθει αυτό σε σύγκρουση με το έργο των εθνικών ε, φορέων για την πιστοποίηση των προσόντων. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικοί φορείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή ε, φέρνουν σε πέρας ε, αυτό το έργο. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ανάλυση του επιδιωκομένου αποτελέσματος και θα πρέπει να υπάρξει και καλύτερο συντονισμός μαζί με τα κρατημέλη να αντλήσουμε κοινά συμπεράσματα για το πώς μπορεί να γίνει η βελτίωση, ο εξυγχρονισμός ώστε για τους εργαζόμενους, για τους φοιτητές, για τους εργοδότες, για τους απλούς πολίτες και τα κράτη-μέλη να μπορεί να είναι εποφελές και χρήσιμο αυτό το έργο και αυτό φυσικά θα πρέπει να περιλάβει και τις, μελλοντικά, ε, τις χώρες που μελλοντικά θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you, ε, Mr. Andrew Lever from ECR. Ευχαριστώ πολύ, Andrew Lever από το ECR, εκ Επιτροπής ε, Πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες Συμπρόεδροι, αυτή είναι μια γενική τοποθέτηση εκ μέρους του ΕΣΥΑΡ. E Θα ήθελα να αναγνωρίσω καταρχάς ε, ότι έχει κάποια σημασία ε, αυτή η πρόταση ε, επειδή από το 2004 έχει ήδη ε, δείξει την αξία του το Europass και για τους χρήστες και για τους νέους αλλά και στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα και ως πριστήν συγκρισιμότητα και αναγνώριζε επίσης και τη σημασία του να δουλεύει δουλεύει κανείς σε ένα πολιτιστικό ε, περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ε, και είναι πολύ σημαντικό το ότι και οι δύο επιτροπές συμμετέχουν στην πρόταση αυτή αναθεώρησης. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να πω ότι το πλαίσιο του Europass ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για τον τελικό χρήστη. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η εθελοντικός του χαρακτήρας και να ε, γίνει σεβαστή η αρχή της αναλογικότητας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και τις ανησυχίες μας, ε, όπως και τους επένους μας για το σύστημα, δεν, δεν ήταν στην αρχή ένα εργαλείο που σκοπό είχε να βοηθήσει στην απόφαση όσων λαμβάνουν αποφάσεις για την απασχόληση, για παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιο έχει την κυριότητα των δεδομένων και ξέρουμε ότι είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ευαίσθητα αυτά τα πράγματα Νομίζω ότι έχουμε εξηγήσει πολλέ φορέ πόσο ευαίσθητοι είμαστε σε θέματα ιδιωτικού βίου των πολιτών και κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή δυστυχώ. Τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορούν να ορίζουν τις δικές τους ομάδες ε, για να μπορούν να συνεργαστούν ε, βάσει της δικής τους εμπεριστατωμένης γνώσης ε, του ακαδημαϊκού τους περιβάλλοντος και η αξιολόγηση πολλών αλληλοεπικαλυπτόμενων εργαλείων όπως το EQF και το ESCO όπως ανέφερε και ο κύριος Μαλίνοφ είναι πάρα πολύ σημαντική ώστε να μην υπάρχει επιπλέον κόστος χωρίς λόγο, ούτε υπερβολική, ε, υπερβολικός φόρτος εργασίας, να υπάρχει διαφάνεια για τους τελικούς χρήστες. Ε, αν άκουσα νομίζω σε μία... Κάποιος είπε ε, ότι μπορεί να υπάρξει μία αναφορά ε, μιας υποχρεωτικής διάστασης αυτού του μέσου. Αν ισχύει αυτό, τότε το ECR θα διαφωνούσε και δεν είναι μόνο η δική μου άποψη αυτή, αλλά και πολλών άλλων συναδέλφων. Καταλαβαίνω λοιπόν το κίνητρο πίσω από την αναθέτηση θεώρηση του πλαισίου ώστε να ε, προσαρμοστεί στι ψηφιακέ δεξιότητε, ώστε να μπορεί το Europass ε, να είναι διαθέσιμο και σε μειονεκτούσες ομάδε. Πράγματι ήταν μια επιτυχής πρωτοβουλία, όμω ένα από του λόγου επιτυχία ήταν ο θελοντικό του χαρακτήρα. Ε, και πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αυτονομία στον τομέα αυτό των κρατών μελών και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζητνάσκα. Έχετε το λόγο. μετά από τον συνάδελφό μου του ECR που αναφέρθηκε και τόνισε ορισμένα σημεία όπως είναι η επικουρικότητα και εγώ θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να διατηρηθεί μεν η επικουρικότητα και πρέπει να πω ότι ναι μεν Χαιρετίζω την πρόταση αυτή, γιατί πράγματι ήταν καιρό να υπάρξει αναθεώρηση του συστήματος του Europass, όπως αναφέρει και η ίδια η πρόταση της Κομισιόν, αυτό το οποίο έχει η πρόταση είναι να εξασφαλίσει ότι θα μπορούν να γίνονται γνωστά τα προσόντα και οι δεξιότητες των ε, ε, εργαζομένων χωρίς να υπησέλθει σε άλλα θέματα <clears throat> όπως είναι η δυνατότητα πληροφόρησης για τις δυνατότητες αυτής της κατάρτισης. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να υπάρξει η προσαρμογή προς τις νέες τεχνολογίες και την διαβίου μάθηση ώστε να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια καλύτερη προσαρμογή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων στις ανάγκες της αγορές. Επίσης όμως θα πρέπει και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναπηρίες όπως χάρη, τα άτομα τα οποία ε, είναι κοφάλαλα, θα πρέπει και αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτονται από αυτό το σύστημα, δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τις πλατφόρμες που δημιουργούνται στα πλαίσια του Europass. Και είναι απαραίτητο επίση να μην υπάρξει υπερβολικό διοικητικό άχθο το οποίο θα συνδέεται με την εφαρμογή αυτού του νέου επικαιροποιημένου συστήματο, Δεν θέλουμε να γίνει αυτό το οποίο συχνά συμβαίνει με τις ε, μεταρρυθμίσεις, δηλαδή να υπάρξει περαιτέρω βάρος και άχθος για τους καταναλωτές, για τους χρήστες και για τα εθνικά κράτη. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Ο κύριος Ιλίαν Καουτσούκ. Δεν είναι παρόν όμως. Λαος Χούντις. Ο κύριος Χούντις ούτε και αυτός είναι παρόν. Ε, Τάνια Γκονσάλες Πένιας. Η Τάνια Γκονσάλες Πένιας ούτε. Τζιλ ε, Evans, όχι. Τομινικ Μπίλντε, ούτε. Okay. Uh, then I give you the word to <laughs> Madam Kammerwert. Ξαναδίνω το λόγο στην κυρία Κάμερβερτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλα μέλη τα οποία ζήτησαν το λόγο, σας παρακαλώ όμως να παραμείνετε σε ένα χρονικό διάστημα ενός με δύο λεπτά. Η κυρία Μονισακή έχει το λόγο. Μονισακή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, διότι το Europass είναι πολύ σημαντικό και αφού έχει περάσει μια δεκαετία υπάρχει περιθώριο για κάποιες διορθώσεις, για μια αναθεώρηση του μηχανισμού αυτού. Τι έχει αλλάξει σε αυτή τη δεκαετία. Έχουμε μια οικονομική κρίση που σάρωσε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και την Ευρώπη με αποτέλεσμα σήμερα υπερβολικά πολλοί νέοι συμπολίτες μας ε, να αναζητούν ε, εργασία. πειραματιζόμενοι σε χώρους όπου υπερβαίνουν ε, την αρχική τους εκπαίδευση ή τη δουλειά που είχαν. Οπότε αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή την αναθεώρηση του Europass είναι να το μπορέσουμε να προσαρμόσουμε το μηχανισμό αυτό ώστε να ε, ενσωματώσει και τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί ε, πέραν του πλαισίου της ε, διαρκούς κατάρτισης ή της αρχικής κατάρτισης. Να ενσωματώσουμε δηλαδή διάφορες δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και αλλού στο σπίτι, σε κάποια, στο πλαίσιο κάποιου οργανισμού, διότι πρέπει οπωσδήποτε τα βιογραφικά του καθενός να εμπλωτιστούν. Οπότε διότι ο απότατο σκοπό είναι να βάλουμε στην αγορά εργασία πολλού συμπολίτε μα. Δεν είναι ένα σύστημα, ένα μηχανισμό που πρέπει να λειτουργεί απλά για να λειτουργεί. Είναι για να εντάξει του συμπολίτε μα στην αγορά εργασία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ε, πολύ καλό το ότι υπάρχει μια ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι έχουν άμεση επαφή με τα τεκτενόμενα. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το μηχανισμό. Ευχαριστώ. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Frau. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σόντροβα, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε πει πολλά για την αναγκή του να υπάρξει μεταρρύθμιση στο Europass. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμα το οποίο λέει και η Κομισιόν και το οποίο το βλέπω να είναι χρήσιμο. Να υπάρξει καλύτερη χρησιμοποίηση του διαδικτυακού, του ψηφιακού συστήματος. Γιατί με τον τρόπο οι... αυτοί που ψάχνουν για εργασία και πρέπει να είναι ορατοί στην αγορά εργασίας γίνονται πραγματικά περισσότερο ορατοί. Τους δίνει με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη ορατότητα, μεγαλύτερη κινητικότητα και δυνατότητα αναγνώρισης των προσόντων τους. Γιατί <clears throat> θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τη μεγαλύτερη χρήση των ψηφιακών συστημάτων. Εδώ πρέπει να εστιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να ενισχυθούν αυτά τα συστήματα. Εγώ θέλω λοιπόν να εστιάσω την προσοχή μου στην μεγαλύτερη ψηφιοποίηση του συστήματο ώστε να προκύψει μεγαλύτερη προσβασιμότητα στο σύστημα. Αυτό δεν οδηγεί προβλήματα στα κρατη Ευχαριστώ, Νέκη πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη, λέει η κυρία Τρούπελ, να αναθεωρήσουμε το Europass. Δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ένα νέο εργαλείο. Θα Πρέπει να αρκεστούμε σε μερικές ε, τροποποίησεις του εργαλείου και συμφωνώ με όσους λένε ότι δεν πρέπει να ρίψω και δεν με την επικουρικότητα όταν τα πράγματα λειτουργούν καλά. Αλλά από την άλλη, όπου βλέπουμε ότι ε, υπάρχει κάποια ανάγκη βελτίωση τη οργάνωση και τη συνεργασία στην Ευρώπη, ε, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, πρέπει οι άνθρωποι να έχουν ευκαιρίες ε, για το μέλλον όσον αφορά τις δεξιότητές τους και να τους αναγνωρίζονται αυτές τις δεξιότητες και οι οριζόντιες δεξιότητες καθώς και οι δεξιότητες κυκλικής και πράσινης οικονομίας. Έτσι υποστηρίζουμε την ανάπτυξη ε, των ε, μελλοντικών τομέων της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας. Οπότε είναι σαφές ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε και να αναπτύξει ο κόσμος και οι ήπιες δεξιότητες. Οπότε πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτές. Θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι άτυπες ε, δεξιότητες. Οπότε κάνουμε έκκληση για ισχυρή υποστήριξη των ε, δραστηριοτήτων επικοινωνίας ώστε να ενημερώσουμε όλους όσοι δεν, δεν ε, συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε όλους τους τρόπους εκμάθησης και παιδείας. Οπότε να μην δείξουμε στενομυαλιά να υπάρξει ευρεία επικοινωνία. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τη, έτσι, την έννοια της απασχολησιμότητας αλλά πρέπει να πάμε πέρα από αυτό, διότι αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε κάτι που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όσον αφορά λοιπόν την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων του προσόντων και τη επαγγελματική εμπειρία μέσω του Eurobus, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι ήπιε και οι άτυπα αποκτηθήσει δεξιότητε θα αναγνωρίζονται. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ε, προσπελασιμότητα στον Europass και την ε, ε, καλύτερη χρήση του από ανθρώπους που βρισκόνται σε ευάλωτη κατάσταση και κάνουμε έκκληση για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, των υπηρεσιών απασχόλησης, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων νέων και των οργανώσεων διαβίου μάθησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νίκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω καταρχήν εξ ονόματος και των συναδέλφων μου της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπορέσουμε να εργαστούμε σε αυτό το θέμα μαζί με τους συναδέλφους της Επιτροπής Απασχόλησης. Οι δεξιότητες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνεκτικές και συνεπείς πολιτικές στα θέματα της παιδείας. Το πρόβλημα της έλλειψης προσόντων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για να μπορέσουμε να μειώσουμε και την υψηλή ανεργία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα της Κομισιόν για τις δεξιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο αναμένουμε εδώ και πολύ καιρό και τονίζει την ανάγκη να υπάρξει και ένα ευρωπαϊκό σύστημα που να έχει κοινά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντα υπόψη και την τωρινή οικονομική συγκυρία. Ένα πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, θα πρέπει να μπορέσουμε να προβλέψουμε τις μελλοντικέ ανάγκες της αγοράς. Δεν είναι οι ίδιες οι δεξιότητες που θα απαιτούνται σε 10, 20, ακόμα και 30 χρόνια με αυτές που χρειαζόμαστε σήμερα. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κατάλληλα στελέχη τα οποία δεν θα είναι μονάχα ικανοί μάνατζερ, αλλά θα είναι και απελευθερωμένοι και ε, ικανή και στα ανθρώπινα ε, διοικητέ επιχειρήσεων και ομάδων. Είναι απαραίτητο λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν κριτικό πνεύμα σκέψης, να έχουν δημιουργικό πνεύμα και να μπορούν να παίρνουν πεφωτισμένες αποφάσεις. Επομένως, μέσα στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να γίνει και μια μεγαλύτερη διάκριση μεταξύ των πραγματικών αντικειμενικών δεδομένων και των ατομικών απόψεων. Μόνο με μια ολιστική άποψη, μόνο με την ανάπτυξη των ικανοτήτων όλων των ανθρώπων, μόνο θέτοντα τον άνθρωπο στο κέντρο αυτού του γίγνεσθε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση λοιπόν στις ε, σπουδές, στην απόκτηση ε, δεξιοτήτων και αυτό να περιλαμβάνει και τα πιο ευάλωτα στοιχεία της κοινωνίας μας, γιατί ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να είμαστε περιεκτικοί, να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα να βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Όσοι δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένοι για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να βοηθηθούν από αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Κομισιόν, λοιπόν, δεν προβλέπει αυτή τη στιγμή κάποιους μηχανισμούς για τον αγώνα κατά της σχολικής αποτυχίας, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένη και θέλω να υπογραμμίσω σχετικά ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 70 εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τις βασικές δεξιότητες, δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάσουν, δεν έχουν ικανότητα να λειτουργήσουν στην αριθμητική και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα συνολικό σύστημα εκπαίδευσης το οποίο αντιμετωπίζει τις κοινωνικές απαιτήσει και έτσι να αντιμετωπίσουμε την σχολική αποτυχία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών μας η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ένα από τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως λέει και η Χάρτα, και οι πολίτες, όλοι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ικανότητες σε όλα αυτά τα θέματα, κυρίως να έχουν και κοινωνικές και ψηφιακές ικανότητες και σε επίπεδο μέσων ε, επικοινωνίας και κυρίως να μπορούν να έχουν την κριτική ικανότητα για να διαχωρίζουν την πραγματικότητα από τις απόψεις. Θα πρέπει εδώ να υπάρξει και μια μεγαλύτερη υπευθυνοποίηση των διδασκόντων και των εργοδοτών. Δυστυχώς, εγώ μιλώντας με διάφορους ανθρώπους, βλέπω ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη κουλτούρα σε επίπεδο εργοδοτών, δεν έχουν την πεποίθηση ότι θα πρέπει να καταρτίζουν σε μόνιμο επίπεδο τους εργαζομένους του. έξω και η σύγκρουση αυτή. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, ενώ οι εργοδότες τους τους λένε κάντε το αυτό, μάθετε ό,τι θέλετε, αλλά όχι την ώρα εργασία. Επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε και για τη δυνατότητα να υπάρχουν ανεξάρτητοι τομεί ε, εκπαίδευση που θα επιτρέπουν την διαβίου αύξηση των ικανοτήτων. Και θέλω επίσης, κλείνοντας, να σταθώ και στους διδάσκοντες. Δεν θέλουμε μονάχα να αυξάνουμε τις τεχνολογικές υποδομές, θα πρέπει να επενδύσουμε και ιδίω μέσα στην κρίση που βρισκόμαστε θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο έμψυχο υλικό των διδασκόντων ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις τεχνολογικές αλλαγές και να συνεχίσουν την σωστή εκπαίδευση των εργαζομένων. Τώρα πρέπει να σταματήσω. Αν θέλετε, στη συνέχεια μπορώ να συμπληρώσω αυτά τα οποία σας είπα για τα θέματα των δεξιοτήτων. Ναι, ναι, βεβαίω μπορείτε να επανέλθετε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Κάμερεφερτ. Ε, θα ήθελα να δώσω τώρα κυρία Μελίντα, λέει η πρόεδρος, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ω σκιώδη εισηγήτρια στην Επιτροπή Απασχόληση θα είχα τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα. Ε, Αυτό ο επιπλέον μηχανισμό ε, θα έπρεπε να διευκρινιστεί ε, γιατί έχουμε έναν γενικό μηχανισμό που αναφέρεται ως ε, ΡΕΣ. Ε, έχουμε επίσης το θέμα των υψηλών, του υψηλού επίπεδου προ, προσόντων που επίσης αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το αναθεωρήσουμε και έχουμε και το σύστημα των προσόντων, το EQF και πρέπει να δούμε πώς συνδέονται όλα αυτά. Η αναθεώρηση 2015 και 2016 δείχνει 27 εκατομμύρια εκατομμύρια επισκέψεις ε, στον ιστότομο, 19 εκατομμύρια ε, βιογραφικά σημειώματα που δημιουργήθηκαν, 58% ε, εκ των οποίων μας λένε οι χρήστες ότι είχε ως αποτέλεσμα μια συνέντευξη ή εκπαίδευση, όμως δεν ξέρουμε πράγματι πόσοι άνθρωποι βρήκαν δουλειά κατά αυτόν τον τρόπο. Επομένως δεν ξέρουμε πολύ καλά αυτοί ε, οι 70 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν, οι 12 εκατομμύρια άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι που έχουν ένα πολύ χαμηλό ε, ποσοστό ε, δεξιοτή, πολύ χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, πώς το χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο. Κατά τα υπόλοιπα υπάρχει μια ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό το βιογραφικό σημείωμα. Δεν, δεν παίζει ρόλο ούτε η εθνικότητα ούτε η χώρα διαμονής, κάτι το οποίο ε, ε, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό ο συνάδελφος Νομινίκ Μπίλντε και εγώ ε, θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς τις ε, διατάξεις που θα υπάρξουν, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας νέος τρόπος μετανάστευσης, για να το πω έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κώστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ τώρα για το Europass, γιατί αυτό εξακολουθούμε να συζητάμε, νομίζω. Αναμφίβολα πρόκειται για μια προσαρμογή ενό εργαλείου που, που έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του μετά από 10-13 χρόνια ζωή. Ωστόσο, πρέπει να προσαρμοστεί στι νέε συνθήκε. Παρότι θεωρώ ότι χρειάζεται ο μέγιστο δυνατό συντονισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά κάποια κράτη-μέλη ανησυχούν ότι μπορεί να υπερφορτωθεί ο μηχανισμός απόψη δαπανών αλλά και διαλειτουργικότητας. Ε, δηλαδή μπορεί να παρεμποδιστεί η εύρυθμη εφαρμογή η οποία ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει ε, εκδιπλωθεί πλήρως. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να υπενθυμίσουμε ότι αν μη τι άλλο θα πρέπει να προσαρμόσουμε το εργαλείο για τρεις ε, λόγους. Πρώτα απ' όλα να ενισχυθούν τα έγγραφα online για όλους ε, και οι υπηρεσίες επίσης και το πώς η ενσωματώση με τα άλλα εργαλεία επίσης, η ολοκλήρωση με τα εργαλεία το ΕΣΚΟ και το ΙΟΡΕΣ. Το ζήτημα του συντονισμού με τα δίκτυα υποστήριξης ε, και η διαλειτουργικότητα. Αυτή είναι φιλόδοξη στόχοι οι οποίοι θα επιτευχθούν σταδιακά, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που έχουν αποκτήσει τεράστια ε, γνώση αυτή τη στιγμή και βοηθούν ε, στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ε, χωρών. Είναι πρόκληση αυτή η πρόοδος του συστήματος που θέλουμε. Τώρα θα πρέπει να αναγνωριστούν πέραν των επίσημων δεξιοτήτων και οι ανεπίσημες, οι άτυπες και έχουμε μαχηθεί εμείς στην Επιτροπή Πολιτισμού για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Έκαρτ από την Κομισιόν. Εάν θέλει βέβαια. Τρία με πέντε λεπτά. Yeah, thank you. Um, uh, what I... Ε, ευχαριστώ αυτό που καταλαβαίνω εγώ από τη συζήτηση αυτή είναι ότι υπάρχει πράγματι μια συνένεση για την ανάγκη ε, εξυγχρονισμού, όπως επίσης και για τη λογική πίσω από αυτή. Τα ερωτήματα αφορούν περισσότερο την κατεύθυνση ε, και πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την αντίδραση των κρατών μελών. Όταν βλέπουμε τις αντιδράσεις των κρατών μελών, μπορώ να ομαδοποιήσω τις ανησυχίες ε, στις εξής κατηγορίες. Παρεξήγηση, έσκο και τρίτον διακυβέρνηση. Και αυτά ήταν τα ζητήματα λίγο πολύ που ετέθησαν και εδώ. Όσον αφορά την παρεξήγηση, ε, πρόκειται για τον χαρακτήρα της απόφασης. Η απόφαση δεν ε, σημαίνει οποιαδήποτε υποχρέωση για τα κράτη-μέλη. Επομένως, όλα όσα υπόθηκαν που αφορούσαν την ε, επικουρικότητα και τη διατήρησή, ε, τη διατήρησή της και κατά πόσο το σύστημα πρέπει να παραμείνει προαιρετικό, αυτό είναι πράγματι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς δεν θέλουμε να προτείνουμε κανέναν υποχρεωτικό χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο. Όταν λέμε για παράδειγμα για τη χρήση του ΕΣΚΟ και του Europass, ε, είναι ε, λογικό. Όταν μιλούμε για το Europass, ε, μιλούμε για, διάφορες, για διάφορα συστήματα ταξινόμησης στα κράτη-μέλη. ΕΣΚΟ θα ήταν το μεταφραστικό εργαλείο που θα χρησιμοποιούσαμε, για να το πω έτσι, όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ελπίζουμε ότι ευρέως θα χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν υπάρχει υποχρέωση να ε, χρησιμοποιήσει κανείς το ΕΣΚΟ. Αυτό νομίζουμε ότι το αποσαφηνίσαμε με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα θα υπάρξει πρόοδος και εδώ. Η αποστολές των 14 κρατών μελών αναφέρθηκαν, ε, ήταν σε επίπεδο επιτετραμένων ε, οι συζητήσεις που έγιναν και έχουν καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά τώρα το ΕΣΚΟ πρόκειται για μια ταξινόμηση και ανείχνευσα από τα σχόλιά σας. Ε, εντάξει, καταρχήν είναι ένα καλό εργαλείο, αυτό είπατε κι εσείς. Το θέμα είναι πώς θα διατυπώσουμε το ε, εργαλείο αυτό στο πλαίσιο της απόφασης. Αυτό ε, είναι η υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή. Και τέλος, η διακυβέρνηση. Είναι όμως εξίσου σημαντική η διακυβέρνηση Έχουμε το Euroguidance, το δίκτυο, το EQF, τα εθνικά σημεία επαφών ε, και ε, τα κέντρα καθοδήγησης για το ε, Europass. Σε μερικές φορές, σε μερικές, μερικές είναι ελεύθεροι οργανισμοί, μερικές φορές συνεργάζονται και αποτελούν τμήμα ενός συστήματος. Η συνεργασία μεταξύ αυτών των δικτύων, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά την ποιότητα της, των μεμονωμένων εργοστασίων, εργασιών, πολλές φορές αυτή η συνεργασία δεν υφίσταται καν. Και αυτό δεν είναι ε, η καλύτερη δυνατή κατάσταση για το μέλλον. Επίση, τα δίκτυα αυτά όλα κρηματοδοτούνται από τον νοσιακό προπολογισμό. Οπότε παρατήρηση δευτερεύουσα σημασία, δεν υπάρχει επιπλέον διοικητικό κόστο. Ε, αυτά όλα καλύπτονται από τον προπολογισμό τη Ένωση. Για αυτά τα τρία δίκτυα έχουμε αρκετά δισεκατομμύρια ε, για, κάθε, ε, για αυτή την προγραμματική περίοδο και το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο πρέπει να ε, συνάψει 110 συμφωνίες επιδότησης. Για μας αυτό ε, δεν είναι μια ε, σωστή ε, διαχείριση του προπολογισμού, γιατί υπάρχει μία υποαξιοποίηση 8 εκατομμυρίων κατέτος. Κατά την άποψή μας, το σύστημα που προτείνουμε θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητα, γιατί θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη ελεύθερα να ε, ε, δίνουν τον προϋπολογισμό αυτό στο σύστημα όπως εκείνα θέλουν. Θα υπήρχε δηλαδή μια καλύτερη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το θεωρούν ευπρόσδεκτο αυτό. Τώρα, ποια είναι η υποχρέωση για τα κράτη-μέλη. Υποχρεώσει για τα κράτη-μέλη είναι οι εξή. Να συμμετέχουν στην πλατφόρμα για τη συνεργασία. Ε, εμείς ε, θα καλύπταμε τα έξοδα όλων των εμπειρογνωμόνων ε, για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα και εξίσου σημαντικό να προωθήσουμε τις προδιαγραφές του Europass. Δεν ζητούμε τίποτε παραπάνω από τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι τα αιτήματά μας είναι αρκετά λογικά θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε τον ε, ε, μελλοντικό χαρακτήρα ε, της πρότασής μας που νομίζω ότι είναι κάτι που το αποδέχεστε γιατί το αναφέρατε κάποιοι στα σχόλιά σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο και στους δύο εισηγητές για να κλείσουμε. Ε, παρακαλώ τήρηστε το χρόνο σας γιατί εμείς θα πρέπει να σταματήσουμε στις 4.30. Ο κύριος Μάν και μετά ο Μάλινοφ. Η διαβίωση ε, παιδεία είναι βασική αρχή για μας και χαίρομαι ότι όλοι συμφωνούν πως δεν πρέπει να είναι το μέσο υποχρεωτικό αλλά ότι είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τον καλύτερο συντονισμό στην καλύτερη συνεργασία, είναι κάτι πολύ σημαντικό και συμφωνώ με αυτό που είπαν οι περισσότεροι ότι αυτές οι ομάδες εμπειρογνωμόνων ε, ήταν αποτελεσματικές. Ε, το έχω σημειώσει και εγώ και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Αλλά ο ρόλος τους πρέπει να παραμείνει κάπως περιορισμένος. Ε, είναι σαφές ότι θα πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικές Ε, έχουμε μια καλή εμπειρία με τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, την οποία πρέπει να συνεχίσουμε. Κάποια πράγματα θα πρέπει να ξεκαθαριστούν φυσικά. Από τα μηνύματα που ακούσαμε ε, θα είναι πολύ βασική η συνεργασία για το μέλλον και χαίρομαι για όλα αυτά που συμφωνήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαλινόφ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Τα πιο σημαντικά τα έχουμε αναφέρει. Υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πράγματι εδώ υπάρχουν προτάσεις που αντιμετωπίζουν τις κέρδες αντιστοιχίες μας. Συνήθως οι εκπρόσωποι των κρατών μελών όταν έχουν κάποιες υποψίες, αντί να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, φαντάζονται τα χειρότερα. Και τότε δημιουργούνται προβλήματα. Όταν είπατε ότι δεν θα υπάρξει υποχρεωτικός χαρακτήρας, αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούσαν καλά τα κράτη-μέλη και ελπίζω ότι μετά από αυτό θα μαλακώσει λιγάκι η θέση τους. Κατά τα άλλα υπάρχει η γενική συνένεση ότι είναι απαραίτητη η, ο απαραίτητος εξυγχρονισμός και αυτό μας δημιουργεί μια βάση για σύνδεσμους. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για αυτή την πρώτη ε, ανταλλαγή απόψεων. 23 Μαρτίου το πρωί θα έχουμε μια περαιτέρω κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Πολιτισμού όπου θα παρουσιαστεί το σχέδιο έκθεση. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 30 Μαρτίου το μεσημέρι στις 12. Η εξέταση των τροπολογιών στις 25 Απριλίου πάλι με μια κοινή συνεδρίαση των δύο εμπλεκομένων επιτροπών και η έγκριση προβλέπεται <clears throat> να λάβει χώρα στις 21-22 Ιουνίου, εάν θέλει ο Θεός. Και θα δούμε μετά πότε θα μπορέσουμε να έρθουμε στην Ολομέλεια. Εν πάση περιπτώσει θα ξανασυνεδριάσουμε ως ε, συνδεόμενες επιτροπές και οι δύο και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της της διάταξης. Και δίνω το λόγο στην πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης. Βεβαίως. 4. Σημείο 4 το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες. Η μεταρρύθμιση του Europass, όπως ξέρετε, είναι μια ψηφίδα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και αυτό είναι ακριβώ το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Η Κομισιό θέλει να ξεκινήσει μια για να εξασφαλίσει ότι η εκπαίδευση για τις δεξιότητες και η υποστήριξη των δεξιοτήτων θα είναι διαθέσιμη σε όλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 70 εκατομμύρια Ευρωπαίων δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να γράφουν και να διαβάζουν. 70 εκατομμύρια. Και ακόμα περισσότερο έχουν χαμηλά επίπεδα αριθμητισμού και ψηφιακές δεξιότητες. Αυτά τους οδηγούν σε αποκλεισμό και ένδια. Πάνω από τους μισούς μακροχρόνια άνεργους που είναι 12 εκατομμύρια θεωρείται <clears throat> ότι έχουν πολύ χαμηλές δεξιότητες. Επομένως αυτό το θεματολόγιο αντιμετωπίζει όλα αυτά τα ζητήματα από το Europass, από το θέμα της επαγγελματικής και ε, ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την κατάρτιση και εκπαίδευση των μεταναστών και των ετούντων ασύρου. Ο στόχος είναι να υπάρξει καλύτερη χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων που είναι διαθέσιμα, να δώσει στους ανθρώπους αυτούς τις νέες δεξιότητες που χρειάζονται και κυρίως τις ψ, ψηφιακές δεξιότητες. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να σας ξαναδώσω το λόγο σε ημάς με ύψιλον πέτρα από την Επιτροπή Πολιτισμού. Και πάλι σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Κάμερεβέτ χωρίς να θέλουμε να επηρεάσουμε και να αμφισβητήσουμε την αρμοδιότητα των κρατών μέλων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, θα πρέπει κατεπηγόντως η Ευρώπη να αντεπεξέλθει στις ε, νέες προκλήσεις, να αντιμετωπίσει τη σχολική αποτυχία, να δώσει την δυνατότητα σε ανθρώπους που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι να έχουν την κατάρτιση και την εκπαίδευση που χρειάζονται και επίσης να προσαρμοστούμε στον κόσμο της ψηφιοποίησης και κυρίως θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων τους εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε υψηλότερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες μας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να σκεφτούμε και τις τυπικές και τις μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης σε ε, επίπεδο διαβίου εκπαίδευσης. Πιστεύουμε λοιπόν ως Επιτροπή Πολιτισμού ότι ο κύριος στόχος της, ε, κατάρτισης, εκπαίδευσης και της κατάρτισης δεν πρέπει να είναι μόνο η απασχόληση, αλλά ότι είναι αυτός σκοπός από μόνη της η παιδεία. Είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η εκπαίδευση για να εξασφαλιστούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διατήρηση των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μεταλλεμπάδευση της γνώσης από γενιά σε γενιά και όχι μόνο εκπαίδευση για την ε, απασχόληση. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν η μεταλαμπάδευση της γνώσης, της κριτικής σκέψης, να υπάρξει δυνατότητα κριτικής ανάπτυξης του πνεύματος όλων των ανθρώπων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανεκτικότητα και δυνατότητα συμβίωσης. Έτσι λοιπόν κάθε άτομο μπορεί να προετοιμαστεί για την κοινωνική ζωή και έτσι θα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσουμε θετικό τρόπο τις αλλαγές <clears throat> στην κοινωνία και στον χώρο της αγοράς και να είναι ενεργοί πολίτες. Είναι γι' αυτό το λόγο απαραίτητο τόσο η Επιτροπή Πολιτισμού όπως και η Επιτροπή Απασχόλησης με το κοινό του έργο να υπογραμμίσουν τη σημασία αυτού του έργου και χαίρομαι πολύ που μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτήν την συζήτηση και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Μαρίζα για να ξεκινήσουμε την εξέταση των δύο εκθέσεων. Uh, Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Τλαμπάγεβα, την εισηγήτρια, όμως δεν είναι εδώ. Ο κύριος Νέκοφ όμως είναι εδώ. Και τώρα θα έχετε το χρόνο που νομίζατε ότι δεν είχατε προηγουμένως όταν πήρατε το λόγο. Uh, you δηλαδή μπορείτε να μιλήσετε εξ ονόματος και των δύο. Τέσσερα-πέντε λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Φτάνει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, συγγνώμη για αυτή την παρεξήγηση, αλλά το Europass είναι ένα από τα δέκα σημεία ε, τα οποία συμπεριλαμβάνει το θεματολόγιο για τις δεξιότητες. Γι' αυτό ε, θα ήθελα να συνοψίσω και αυτά που είπα και προηγουμένω, ότι οι σημερινέ ε, που είναι, οι σημερινές δεξιότητες που είναι απαραίτητε σήμερα δηλαδή, δεν είναι αυτέ υποχρεωτικά που θα χρειαζόμαστε στο μέλλον. Οπότε πρέπει στο επίκεντρο ε, ο σπουδαστή, ο φοιτητή να, να, πρέπει να είναι στο επίκεντρο τη προσπάθεια ο σπουδαστή, ο φοιτητή για να μπορέσει να αποκτήσει δεξιότητε, που θα του είναι χρήσιμε και απαραίτητες στο μέλλον. Για παράδειγμα, Ε, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να διακρίνει κανείς ε, τα γεγονότα από τις ε, απόψεις, όπως επίσης και από την ευθύνη η καταπολέμηση της εγκατάλειψης του σχολείου. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε ότι 70 εκατομμύρια άνθρωποι ε, στην Ευρώπη δεν ε, ε, έχουν επαρκείς δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταπολεμήσουμε εξαπαλώνων ήχων από την παιδική ηλικία και πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουμε για ε, το μέλλον ε, και να δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή ε, σε αυτήν την πρωτοβουλία των των ε, οδών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, upskilling pathways, ε, ειδικότερα όσον αφορά το χαμηλό επίπεδο ε, δεξιοτήτων και πώς μπορούν αυτές να αναβαθμιστούν. Και μιλάω και για τις άτυπες, και για τα άτυπα προσόντα. Πρέπει να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αυτή τη διαδικασία Πιστοποίηση των δεξιοτήτων, ε, γιατί μπορεί να χρειάζεται χρηματοδότηση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν σταματάει αυτή η χρηματοδότηση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για να αποκρισταλώσουμε όλα αυτά που έχουμε επιτύχει και να πιστοποιούνται αυτές οι άτυπα αποκτηθήσεις ε, δεξιότητες. Ε, αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε αυτό ε, το πρόγραμμα ε, ε, πιστοποίησης των άτυπων προσόντων να αναπτυχθεί. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλούμε πολύ για ψηφιακές δεξιότητες όπως επίσης και για ε, τις δεξιότητες στο πλαίσιο του επιχειρήν. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί να προσέξουμε λίγο με αυτό το μύθο, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο δεν αλλάζει ε, το είδος των δεξιοτήτων μετά την κρίση και λόγω αυτής της κρίσης. Έχουμε μειώσει τις ε, ε, επιδοτήσεις για τους διδάσκοντες στα σχολεία και αυτό δεν βοηθά πολύ την κατάσταση γιατί δεν έχουμε πλέον ικανούς διδάσκοντες που να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση. και μιλάω και για το STEM ε, και τις ε, δεξιότητες ε, που συμπεριλαμβάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι διδάσκοντες να μπορούν να μεταφέρουν αυτή τη γνώση σε κάθε ηλικία για να μπορέσουν μετά ως άνθρωποι να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Πρέπει επίσης να ε, ενισχύσουμε ε, το πόσο ελκυστική είναι η επαγγελματική κατάρτιση. Και αυτό ε, χρειάζεται ένα επίπεδο γνώσεων και πρέπει να ενισχύσουμε ε, τις ε, επαγγελματικές δεξιότητες, δηλαδή να μπορούν τα παιδιά να μάθουν ένα επάγγελμα στο σχολείο. Και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ένα μέλλον στους ε, φοιτητές, που, στους μαθητές που μετά τα 19 δεν θέλουν να σπουδάσουν άλλο και θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό, η ποιότητα και η ποσότητα των ε, διδασκόντων ε, πρέπει να είναι η κατάλληλη, ακόμη και στις αραιοκατοικημένες περιοχές. Πρέπει να ε, βελτιώσουμε τις ικανότητες και τα προσόντα των διδασκόντων. Ένα πακέτο πολλαπλών μέτρων για παράδειγμα την ε, ε, άτυπη εκπαίδευση, την ε, εξατομικευμένη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, μία πρώιμη εκπαίδευση για τα παιδιά, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά αυτά, ακόμη κι αν οι απαιτήσει αλλάξουν σε 10 χρόνια. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο και να, να δώσω το λόγο και στον σκιώδη εισηγητή. Ε, να αναφέρω όμως και κάποια πράγματα εκ μέρους της συνεισηγήτριας της κυρίας Ντλαμπάγιοβα. Επιτρέψτε μου να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της για την απουσία της. Θα ήθελε λοιπόν να τονίσει την, ε, το θέμα της πρόβλεψης των μελλοντικών δεξιοτήτων. Όσον αφορά τώρα την ε, πρακτική ενημέρωση, όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση που ανέφερα προηγουμένως, συμφωνεί και εκείνη, σύμφωνα με την κυρία Ντλαμπάγιοβα, ε, η πρακτική εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης και επίσης πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την επιχειρηματικότητα. Είναι μια, ε, είναι μια διαβίου μάθηση αυτή, ε, είναι υπέρ της διαβίου εξέλιξης ε, του εργαζομένου. Οπότε η κυρία Τλεμπάγεβα συμφωνεί ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση για να καταπολεμήσουμε και την ανεργία. Με πολύ χαρά αναμένει τη συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. You, Ευχαριστούμε ο κύριος Νέκοφ μίλησε επίσης και εκ μέρους της κυρίας Ντλαμπάεβα. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Σόιντροβα. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω τώρα ως η ε, εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚΑ και θα σας μιλήσω για το ε, νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Ε, με ικανοποιεί η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η οποία είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη, περίπλοκη και εστιαστέ στις δεξιότητες, κάτι αποφασιστικό για την ανάπτυξη και την αποσχολησιμότητα στην Ευρώπη. Ε, ενισχύουν το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης, κάτι που είναι ο βασικός σκοπός αυτού του θεματολογίου και πιστεύω ότι κινούμαστε σωστά. Είναι σωστός ο στόχος αυτός. Το θεματολόγιο βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Αναφέρατε 70 εκατομμύρια πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση. Και θέλω να πιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα φτάσουν ποτέ στη δευτεροβάθμια ε, εκπαίδευση, ωστόσο είναι ορατός ο κίνδυνος αυτός ε, και με τον κίνδυνο του να μην μπορούν να αποσχοληθούν πουθενά. Ε, το πρώτο εργαλείο, η εγγύηση των ε, δεξιοτήτων, αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα αυτό τον κίνδυνο και χαίρομαι που το πρώτο αυτό εργαλείο αποτελεί την εγγύηση απόκτησης δεξιοτήτων. Ε, πολύ καλή αυτή η ιδέα της Κομισιόν, διότι όταν δεν έχει κάποιος ούτε τις βασικές δεξιότητες, η απασχολησιμότητά του στο μέλλον είναι πολύ πιο δύσκολη. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι νέο που δεν μπόρεσε να συμπεριλάβει η Κομισιόν, διότι είναι κάτι που συνέβη τον περασμένο Δεκέμβριο. Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του ΠΙΣΑ 2015 και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει επιδείνωση κατά μέσο όρο. Μιλήστε για 70 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς τις βασικές δεξιότητες. Ωστόσο, εγώ έχω να πω ότι η πραγματική αριθμή πρέπει να είναι ακόμη χειρότερη, Διότι δυστυχώς όλο και περισσότεροι μαθητές ε, στην ηλικία των 15 εξακολουθούν να μην έχουν τις βασικές ικανότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα στόχο 15% εκεί να μειωθεί, ο να μειωθεί κατά 15% ο αριθμός των νέων ανθρώπων χωρίς τις βασικές δεξιότητες και αυτή τη στιγμή στο 15%, ε, ε, στο 15 θέλει να το μειώσει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 20% ή και στο 30%. Οπότε, σωστό, δικαίωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει αυτό το θέμα. Δεύτερο εργαλείο είναι η αναθεώρηση των βασικών δεξιοτήτων και εδώ συμφωνώ. Η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς ε, του Εργαλείου 4, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων. Έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό. Μετά έχουμε το εργαλείο των προφίλ των επικών τρίτων χωρών, κάτι που σχετίζεται με τη μετανάστευση, το 7, το Europass και το 8, την καταπολέμηση της διαρροής εγκεφάλων. Ε, και ε, ούτε εδώ προτείνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορούν κιόλα για να είμαστε ειλικρινεί. Πρέπει να δούμε κατά μετά το γεγονό ότι η διαρροή εγκεφάλων αποτελεί τεράστιο πρόβλημα το brain drain ε, όχι μόνο από μια χώρα σε μια άλλη, αλλά και εντό των ίδιων χωρών. Οπότε η καταπολέμηση του προβλήματο τη διαφύγης εγκεφάλων αποτελεί ε, καθήκον όχι μόνο της Κομισιόν, αλλά και των κρατών μελών. Μετά έχουμε το εργαλείο αριθμό 9, την τομεακή συνεργασία και το 10 ε, παρακολούθηση. των ε, πτυχίουχων ε, ε, πανεπιστημιακών πτυχίων. Το ζήτημα είναι τι κάνουν μετά από την αποφύτισή τους, ποια, πόσο αποτελεσματική είναι η τριτοβαθμία εκπαίδευση, γιατί και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως στόχο το 40% του πληθυσμού να έχουν πανεπιστημιακά πτυχία. Εγώ βλέπω τα πλέον εκτίματα της πρώτης, το ότι στοχεύει σε συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά διαβλέπω και κινδύνους. Ε, όπως ανέφερα έχουμε 10 εργαλεία και ο βασικός κίνδυνος είναι ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξη η πρόταση αυτή. Αν μπορούσαμε να εστιαστούμε μόνο σε λιγότερους βασικούς στόχους θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Αλλά το φάσμα των θεματών είναι τόσο ευρύ που πιστεύω ότι είναι ανέφικτο να επιτευχθούμε στο 2020. Συμφωνώ με, τις βασικέ, με τους βασικούς προσανατολισμούς, απλά θεωρώ ότι η υλοποίηση όλων αυτών αποτελεσματικά δεν είναι κάτι ρεαλιστικό. Εγώ λοιπόν θα προτείνω στο μέλλον να ε, ε, περιορίσουμε το εύρος ε, και υπάρχουν και κάποια πράγματα που μου αρέσουν στο θεματολόγιο εστίασης στους διδάσκοντες διότι για να αυξηθούν οι δεξιότητες να βελτιωθούν οι δεξιότητες και, να εστιαστούμε, και για να εστιαστούμε στην απασχολησιμότητα κατά την αναθεώρηση των βασικών ε, δεξιοτήτων. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει χωρίς διδάσκοντες. Μεταξύ των 10 λοιπόν εργαλείων, ε, προλαμβάνω των 10 αυτών εργαλείων, δεν βλέπουμε κανένα από αυτά να εστιάζεται στους διδάσκοντες και αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Φυσικά πρέπει να πω απαραίτητο ότι το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων Ε, δεν εξαλειφθεί όλα όσα είχε προτείνει παλιότερα στην, ε, στο θεματολόγιο εκπαίδευση και παιδεία κομισιών ε, παιδεία και κατάρτιση, συγγνώμη. Και εκεί δίνονταν κάποια προσοχή στου διδάσκοντε. αλλά ένα νέο θεματολόγιο για τι δεξιότητε χωρί να υπάρχει υποστήριξη για του διδάσκοντε, πιστεύω ότι είναι λάθο ω απόφαση. Σα ευχαριστώ και αντιλαμβάνομαι πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα βέβαια. Ευχαριστώ. Για να δούμε τώρα, Εμίλιαν Πάβελ δεν είναι εδώ. Εμίλιαν Παβέλ, ούτε κάποιος αντικαταστάτης του, ε, ούτε ο κ. Λέολ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ECR υποστηρίζει πάντα τις δράσεις οι οποίες οδηγούν σε οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και φυσικά εμπλέκεται και εδώ η εκπαίδευση. Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη σοβαρότερα την σύνδεση μεταξύ διαξιοτήτων και αγοράς εργασίας. Η Κομισιόν μπορεί να έχει κάποιες προτάσεις, αλλά η επικουρικότητα, η τοπική γνώση της αγοράς και των ε, χασμάτων που υπάρχουν σε εκπαίδευση και κατάρτιση είναι σημαντική. Πρέπει να ξέρει κανείς για ποιους αναφέρεται και ποιοι είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι το αντικείμενο αυτών των ε, προγραμμάτων. Είναι καλύτερο λοιπόν από το να έχουμε μεγαλώσιμα σχέδια να κάνουμε αυτό το οποίο είναι το απαραίτητο. Χωρίς μια ενιαία στάση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν είμαστε κάπως σκεπτικιστές σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Δεν θέλουμε να υπάρξει κεντρική χρηματοδότηση από, ε, από ένα χώρο που υπάρχουν ήδη πολλές, πολλοί περιορισμοί στην ε, χρηματοδότηση. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπερφορτώσουμε με κόστος την ε, εκπαίδευση και όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι είναι απαραίτητο να εστιάσουμε καλύτερα σε αυτήν την ε, έκθεση και αυτό θα είναι και ο στόχος του ECR. Σας ευχαριστώ. Και αν Κουτσούκ δεν είναι εδώ, δεν είναι και ο επόμενος συζήτης. Η Χέλγα Τρούπελ. θα μιλήσει εξ ονόματος των Πρασίνων. Έχετε το λόγο. Επανέλθω στο σημείο αυτό το οποίο είχε να κάνει με τη μεταρρύθμιση του Europass. Επομένως, το ερώτημα είναι ποια είναι η δική μας αντίληψη για την εκπαίδευση. <clears throat> Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εκπαίδευση για την απασχόληση. Θα να υπογραμμίσω και πάλι αυτά που είπε η πρόεδρο τη Επιτροπή μα, ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε μια αντιμετώπιση που βασίζεται μονάχα στην απασχολησιμότητα. Εμεί ω Επιτροπή ε, κουλτούρα θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εκπαίδευση και για το μέλλον της κοινωνίας μας και όχι μονάχα για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι είναι ιδιαίτερο να σκεφτούμε και τις ήπιες δεξιότητες, την άτυπη εκπαίδευση των ανθρώπων, να σκεφτούμε τα εκατομμύρια αυτά που δεν έχουν ε, την ικανότητα να γράφουν και να διαβάζουν ή να χειρίζονται αριθμούς, όλα αυτά τα άτομα θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβαση σε μια άτυπη εκπαίδευση και αυτό θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην, ε, στο θεματολόγιο μας για τις νέες δεξιότητες θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε την ενσωμάτωση των ατόμων αυτών ώστε να δώσουμε νέες ευκαιρίες στους νέους οι οποίοι βρίσκονται σε αντίξωες και δύσκολες συνθήκες και επομένως αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και για το Europass και για την απόκτηση νέων ε, δεξιοτήτων και το θεματολόγιο αυτό. Ο κύριο, η κυρία Νταμάτο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που λαμβάνουν χώρα ταχύες αλλαγές, <clears throat> ιδίω σε περιοχές που έχουν υποστεί τα αποτελέσματα της κρίσης και της λιτότητας, η πρόταση για ένα νέο θεματολόγιο για τις ε, ταξιότητες μπορεί να βοηθήσει την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασία πρέπει να ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντα επικυροποίηση των ε, στοιχείων και της ε, δεξιότητας των ανθρώπων σε μια ρευστή αγορά και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αυξήσουμε και την απασχόληση αλλά να αυξήσουμε και την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Οι προτάσεις λοιπόν της Κομισιόν για ένα ελάχιστο επίπεδο δεξιοτήτων και για μια συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πολύ σημαντικό γιατί σε πάρα πολλές περιοχές μα, της Ευρώπης βλέπουμε να αυξάνεται ο αναλφαβητισμός. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε ιδιαίτερα στα στοιχεία αυτά. Θα πρέπει να αποφύγουμε η, η εκπαίδευση, η κατάρτιση να διέπεται από άχρηστες και περιττές πρωτοβουλίες, όπως πολλές φορές βλέπω στη δική μου χώρα, στην Ιταλία. Επίσης, δεν πρέπει να αναχθεί αυτή η προσπάθεια σε ένα εγχείρημα μονάχα ε, προπαγάνδας. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα καταμέτρησης της επιτυχίας στον τομέα αυτό. Υπάρχουν πολλά εκατομμύρια πολιτών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν αυτή τη πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Μπίλντα δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μαρτάν θέλει να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα. Οπότε δίνω το λόγο και πάλι στην κυρία Κάμερεβέρτ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαν με δύο με την αίτηση αν μπορεί σε ένα λεπτό να λάβει το λόγο γιατί αλλιώς έχουμε καθυστερήσει κύριε Μαν. Εγώ θα προσπαθήσω να εστιάσω στα θέματα αυτά. Η κυρία Τρίπελ και η πρόεδρος τόνισαν στο ότι πρέπει να σταθούμε στο θέμα της, ε, της ε, αντίληψης εκπαίδευσης. Έχουμε όμως αποκομίσει μια μεγάλη ε, πείρα ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ της καθαρής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην ε, απόκτηση μιας θέσης απασχόλησης. Υπάρχει το θέμα όμως το οποίο θέλω να σταθώ της σχολικής αποτυχίας. Φεύγουν πολλοί από το σχολείο για να βρουν μια δουλειά. Αλλά αυτό ουσιαστικά σε φέρνει στο χειρότερο όλων των δυνατών κόσμων. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν αυτούς τους νέους οι οποίοι βγαίνουν μετά στην αγορά εργασία με ελληματικά προσόντα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια καλύτερη σύνδεση του σχολείου και της απασχόλησης ώστε να δώσουμε τις απαραίτητες ευκαιρίες στους νέους, να τους δώσουμε κίνητρα ώστε ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το σχολείο να μπορέσουν να επωφελθούν από τις ευκαιρίες γιατί πολλέ φορέ έχουμε παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειε που δεν δίνουν διάρα για τη σχολική εκπαίδευση και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ένα λεπτό λοιπόν, εντάξει. Ναι, ναι. Κοσλόφσκα. Κύριε Κοσλόφσκα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, Καταρχά θα ήθελα να πω ότι αυτό το θεματολόγιο είναι πολύ ευπρόσδεκτο. Υπάρχει ένα συσχετισμός μεταξύ τη αγορά εργασία και και ε, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, ε, της εκπαίδευσης. Υπάρχει μια ε, σφαιρική προσέγγιση. Αυτό το έγγραφο διατυπώνει μία υπόθεση. Δηλαδή, αν υποθέσει κανείς ότι ε, ο, οι δεξιότητες είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει κανείς ε, με εξωτερικό τρόπο. Όμως δεν αρκεί να έχει κανείς ε, επαρκή και πολλά σχολεία, αλλά πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα οι άνθρωποι ε, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος να μπορούν να λάβουν αυτές τις ε, ε, γνώσεις. Πρέπει να σκεφτούμε για παράδειγμα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που μπορούν να εμπλουτίσουν την ε, το, το, την αγορά εργασίας μας. Στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του ποσοστού των ατόμων ε, που έχουν βασικές δεξιότητες χαμηλού επίπεδου και τις ε, πολύ υψηλού επίπεδου δεξιότητες. Από τη μία χώρα στην άλλη είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάντοτε υπάρχει ε, ένα ποσοστό ανθρώπων σε κάθε χώρα που έχει περάσει από τη βασική εκπαίδευση αλλά δεν έχει αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκάρτ από την Κομισιόν έχει το λόγο. Σας παρακαλώ κάντε ό,τι μπορείτε για να είστε σύντομος. <laughs> Έχετε το λόγο κύριε Εκάρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μπορώ να το κάνω. Δύο παρατηρήσεις, δύο ομάδες παρατηρήσεων μάλλον. Η πρώτη ομάδα αφορά τη λογική του θεματολογίου δεξιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίτηδες επικεντρώνεται σε αυτή την περίπτωση στην απασχολησιμότητα. Αυτό ήταν μια σαφής επιλογή. Δεν θέλουμε να παραγνωρίσουμε την ευρύτερη σημασία της διαβίου μάθησης, της εκπαίδευσης για τους πολίτες κλπ όμως ε, υπάρχει μια διεξοδική συνεργασία ε, μέσω της ε, διακήρυξης των Παρισίων, για παράδειγμα, που αναφέρατε. Δεν χρειάζεται στο θεματολόγιο για τις δεξιότητες να επαναλαμβάνουμε πράγματα που έχουμε καλύψει αλλού. Εφόσον υπάρχουν ήδη, υπάρχουν ήδη το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, έκανε μια πρόταση για τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης. έχουμε στόχους στο πλαίσιο της στρατηγικής το 2020. Ε, δεν θέλουμε όλα αυτά λοιπόν που έχουμε καλύψει αλλού να τα επαναλάβουμε, γι' αυτό επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στο ζήτημα τη απασχολησιμότητα, γιατί ήταν ένα λιθαράκι που έλειπε στη στρατηγική μα για να υπάρχει μια σχέση μεταξύ τη ανεργία των νέων, για παράδειγμα, και τη εκπαίδευση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να τονίσουμε στο πλαίσιο του θεματολογίου δεξιοτήτων, ειδικότερα για του νέου, Προσπαθούμε να δούμε Συγκεκριμένε ομάδες όπως για παράδειγμα τα 70 εκατομμύρια ανθρώπων που αναφέρατε. Προσπαθούμε λοιπόν να εντοπίσουμε συγκεκριμένες ε, ομάδες ε, που παρουσιάζουν πρόβλημα και να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένα νέο στοιχείο στο θεματολόγιο που είναι η έντονη συμμετοχή των εργοδοτών. Οι εργοδότες δηλαδή να συμμετέχουν περισσότερο στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. Και αυτό με οδηγεί στη δεύτερη μου ε, ομάδα παρατηρήσεων ε, που αφορά τη σημασία του θεματολογίου αυτού για το μέλλον. Πολλοί αναφέρονται στην τρίτη ή τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, κάποιοι αναφέρονται ε, στο βιομηχανία 4.0, άλλοι λέγονται ότι είναι απλώς ε, μία νέα κατάσταση για το μέλλον που πρέπει να προβλέψουμε είναι γεγονός ότι ε, το εργασιακό περιβάλλον θα αλλάξει άρδιν και πρέπει πολύ περισσότερο να επενδύσουμε στο ε, εργατικό δυναμικό μας και στο εκολαπτώμενο εργατικό μας δυναμικό, δηλαδή τους νέους. Πρέπει λοιπόν να το συνδέσουμε αυτό και με διεθνή φόρα, από συζήτηση για παράδειγμα των G20 στον Ταβός, το θέμα της επένδυσης στις δεξιότητες είναι ένας θεμέλιος λίθος για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ε, που θα ε, προκύψουν από τις ε, αλλαγές που θα επέλθουν. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για όλα αυτά τα σχόλια και τις συστάσεις για το πού πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Έκαρτ. Και ένα λεπτό εισηγητής, αλλά όχι παραπάνω από ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πέτρα. Νομίζω ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το οποίο έμαθα από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι η Κομισιόν θέλει να πετύχει τον ίδιο στόχο με μας. Να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή και από την πλευρά των εργοδοτών για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο τις ε, δεξιότητες που θα αποκτήσει ο εργασόμενος γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ψηφιακή επανάσταση, να δούμε ποιε είναι οι δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητε για να βρει μια νέα δουλειά. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στο άτομο για να μπορούμε να έχουμε την πρέπουσα επαγγελματική κατάρτιση και να υπάρξει μια, ένας διτός χαρακτήρας στην εκπαίδευσή του, ώστε να έχουμε άτομα τα οποία όχι μονάχα ε, θα μπορούν να βρουν μια δουλειά, αλλά θα έχουν και τις απαραίτητες δεξιότητες και την προετοιμασία να αντιμετωπίσουν τις αραγές του μέλλοντος. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να τονιστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αναφέρεται στην έκθεση αυτή. Θα πρέπει να σκεφτούμε και περισσότερο, όπως ο κύριος Τουμάν, για το θέμα της σχολικής ε, αποτυχίας, για να αποφύγουμε να έχουμε αυτά τα 70 εκατομμύρια που δεν μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν ούτε να υπολογίζουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Κάμερεβερ. Νομίζω ότι και για τις δύο επιτροπές μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Σας υπενθυμίζω το, τον οδικό μας χάρτη. 23 Μαρτίου το πρωί θα έχουμε και πάλι μια κίνη ε, συνεδρίαση όπου θα εξετάσουμε και τις τροπολογίες στις, ε, στη συνέχεια 25 Απριλίου και πάλι σε μια δεύτερη κίνη μας συνεδρίαση και η λήψη απόφασης θα γίνει στις 21-22 του Ιουνίου. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτή την έκθεση στην Ολομέλεια, αλλά θα το δούμε όταν έχουμε διεκπαιρεώσει την κοινή ψηφοφορία. Και μπορώ να ξαναδώσω τώρα το λόγο στη Μαρίζα. Ευχαριστώ, Πέτρα. Θα γίνουν και άλλες συνεδριάσεις ε, ε κοινέ μεταξύ των επιτροπών μας. Η επόμενη κοινή συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 23 Μαρτίου από τις 9 μέχρι τις 10.30 το πρωί. Σας ευχαριστώ όλους. Ας περάσουμε τώρα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης. Όποιοι επιθυμείτε να παραμείνετε και να μας ακούσετε, φυσικά είστε ευπρόσδεκτοι. Μια σύντομη ανακοίνωση για τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού. Είναι ελεύθερα, αλλά οι συντονιστές έχουν συνεδρίαση στο PHS 4β. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνεδρίαση. And we who stays here on the... Λοιπόν, και όποιοι μείνουν εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης, περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Είχαμε κάποια αλλαγή της σειράς των θεμάτων. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013-2017 και παράτασή του για την περίοδο 2018-2020. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Να δώσουμε λίγο χρόνο σε όσους φεύγουν ένα λεπτό και μετά θα συνεχίσουμε με το σημείο 7.